Ladies and gentlemen, we are few Κυρίες και κύριοι, έχουμε καθυστερήσει λίγα λεπτά. Ας ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της συνεδρίασης της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Θα έχουμε μια δημόσια ακρόαση για ένα πολύ σημαντικό ε, θέμα, την θαλάσσια διάσταση της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Καλωσορίζουμε τη συνάδελφο Ανά Γκόνμες, η οποία συντάσσει τη σχετική έκθεση και σίγουρα θα έχετε πολλές ερωτήσεις για τους ομιλητές μας. Έχουμε τρεις διακεκριμένους προσκεκλημένους. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Χιού Γκρίφιθς από το Ερευνητικό Ινστιτούτο της Στοκχόλμης για τη Διεθνή Ειρήνη, τον ε, δόκτορα Τιάγκο Πίτα Εκούνια, δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομά σας, σύμβουλο θαλασσίων υποθέσεων ε, του Προέδρου της Πορτογουλίας και τον αντινάβαρχο αναποστρατεία Λουτς Φέλτ, πρώην αρχηγό του Γερμανικού Ναυτικού. Να, να ζητήσω καταρχάς από τον κύριο Κρίφης να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Νομίζω ότι θα έχετε 15 λεπτά ο καθένας. Το γνωρίζετε αυτό και θα έχουμε και ε, χρόνο για ερωτήσεις. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Εκ μέρους του Ερευνητικού Ινστιτούτου της Στοκχόλμης για την Ειρήνη Διεθνώς, καλωσορίζουμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται να συνεισφέρουμε και εμείς στη συζήτηση για τη στρατηγική για τη θαλάσσια ασφάλεια και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό στο οποίο δεν δίδεται συχνά η σημασία που του αξίζει. Να σας δώσω κάποια στοιχεία για την βιβλιογραφία στην οποία έχει καταλήξει το Ινστιτούτο μας. Μία πρώτη μελέτη για την ευρωπαϊκή διάσταση έγινε μετά από αίτημα του Γαλλικού Υπουργείου Αμήνης και στη, διαφάνεια βλέπετε το εξώφυλλο η λύση που βρήκαμε για αυτό το ε, θέμα ε, έχει καθαρά ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Το 2009 και το 2010 είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με πολλούς εμπειρογνώμονες, τον αντινάβαρχο Λούτς Φέλτς και τον, ε, την Σοφή του Πένα, και καταλήξαμε σε μηχανισμούς που μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο για την ασφάλεια της ναυσιπολίας. Έχουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ΕΜΣΑ, έχουμε τις διάφορες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλους τους άλλους παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτό το τομέα. Με αυτή την πρώτη μελέτη κατανοήσαμε πολύ καλά τόσο το εξαιρετικό έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή, αλλά και όσο και τις προκλήσεις ε, που κρύβονται πίσω από την ε, προώθηση προς το μέλλον αυτής της στρατηγικής. Η έκθεση για το Γαλλικό Υπουργείο Αμήνης δεν είναι δημοσιεύσιμη. Μπορώ όμως να σας δώσω τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αξιωματούχων του Γαλλικού Υπουργείου Αμήνης και μπορείτε να το ζητήσετε αντίγραφο και μπορείτε από τη διαδικτυακή μας ιστοσελίδα να κατεβάσετε, να φορτώσετε το έγγραφο πολιτικής του Ινστιτούτου μας, του ΣΥΠΡΙ. Και είναι η πρώτη φορά που περιλαμβάνεται σε μία έκθεση ανοιχτή για όλους στοιχείο που έχει να κάνει με τα πλοία που εμπλέκονται στην, στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Είναι η έκθεση αρκετά πυκνή και έχουμε πάρα πολλά στοιχεία εκεί και τα οποία αντλούμε από την VIMIT που είναι η βάση δεδομένων για τα συμβάντα με σκάφη και για τα συμβάντα στην ναυσιπλοεία. Είναι μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει 2.500 συμβάντα αλλά και ε, εκθέσεις που έχουν να κάνουν με 15.000 πλοία ή σκάφη. Περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η σημαία του πλοίου, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα δρομολόγια, θέματα ασφάλειας, ρήπανσης αλλά και συγκρούσεων. Θα ήθελα συνοπτικά να σας αναφέρω τα βασικά ευρήματα της έκθεσης που δεν θα σας εκπλήξουν πιστεύω. Πρώτον, οι μεταφορές οι θαλάσσιες κυριαρχούν στο λαθρεμπόριο τόσο παράνομων αγαθών αλλά και στο εμπόριο νομίμων αγαθών. Είναι σαφές ότι η μεταφορά διαθαλάσσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο λαθρεμπόριο ναρκωτικών και στις σχετικές ροές των χημικών πρόδρομων ουσιών. Έχουμε ε, την πλειοψηφία του λαθρεμπορίου καπνού, ε, πετρελαίου αλλά και παραποιημένων ε, εμπορικών προϊόντων η οποία μεταφέρεται δια της θαλάσσιας οδού αλλά και οι περισσότερες δεσμεύσεις, κατασχεύσεις και παρακολουθήσεις ύποπτων φορτίων στρατητικού εξοπλισμού αλλά και προϊόντων διπλής χρήσης γίνονται δια θαλάσσης και προέρχονται ή προορίζονται, προέρχονται από ή προορίζονται προς το Ιράν μεταξύ άλλων. Έχουμε εδώ, την, ε, βλέπετε εδώ τα σκάφη και τα πλοία κατηγορίας 1 ε, της πρώτης κατηγορίας. Ε, είναι αυτά που εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή όπλων και τον οποίων ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ή αυτός που τα λειτουργεί εν πάση περιπτώσει εμπλέκεται σε αυτό. Η περίοδος είναι από το 1991 μέχρι το 2011. Στην μπλε στήλη βλέπετε το ποσοστό που καταλαμβάνουν αυτά τα πλοία στο συνολικό στόλο εμπορικής ναυτιλίας από το 1991 μέχρι το 2011. Στην κόκκινη στήλη βλέπετε το ποσοστό ε, που καταλαμβάνουν στη βάση δεδομένων του ΣΥΠΡΙ, του Ινστιτούτου μας στη Στοκχόλμη. Ο Παναμάς, όπως γνωρίζετε, είναι η χώρα ε, της οποίας τη σημαία επιλέγουν τα περισσότερα σκάφη και πλοία στον κόσμο. Επομένως υπάρχει μεγαλύτερη αναλογία, αντιστοίχως. Και μάλιστα, ε, ίσως εδώ πέρα βλέπετε ότι τα πλοία με σημαία Παναμά μας εκπλήσουν, γιατί δεν είναι παρόντα σε μεγάλο βαθμό. Ε, και αυτό φαίνεται ακόμα περισσότερο στην περίπτωση της Βόρειας Κορέας. Εκτός από το Ιράν και την Κίνα, όλες, όλα τα κράτη που βλέπουμε τη σημαία τους εδώ είναι ανοιχτού μητρώου, όπως το λέμε, ανοιχτού νιολογίου, δηλαδή σημαίες ευκαιρίας. Και εκεί οι κανονισμοί για την ασφάλεια ε, τείνουν να εφαρμόζονται λιγότερο ε, συγκριτικά με τις άλλες χώρες. Βλέπετε λοιπόν ότι ο βαθμός απορρίθμησης είναι πολύ υψηλός και αυτή η τάση διαφαίνεται συνεχώς στην έκθεσή μας ως προς την, ε, το καθεστώς δικαιοδοσίας των χωρών αυτών στον οποίο τον να είναι εγγεγραμμένα αυτά τα πλοία. Επομένως, ο κανονισμός για την ασφάλεια είναι ε, καθοριστικός. Και θα ήθελα να σας δείξω μια διαφάνεια για αυτό το οποίο ονομάζουμε PSC, Port State Control, έλεγχος ε, ε, λιμένων και είναι κάτι το οποίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται πολύ καλά. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προσχωρήσει στο μνημόνιο των Παρισίων για τον έλεγχο των ε, ε, λιμενικών αρχών η Γενική Διεύθυνση ΜΟΥΒ αλλά και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας εργάζονται και είναι πολύ αποτελεσματικοί στη δουλειά τους. Έχουμε ε, μαύρες ε, λίστες ε, των κρατών που προσφέρουν σημαίες ευκαιρίες και που δεν έχουν καλές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια. Αλλά και στη ΣΥΠΑ έχουμε την ακτοφυλακή των ΗΠΑ που κάνει επιθεωρήσεις, ελέγχους και αποτελεί το αντίστοιχο για, συνεισφέροντας σε αυτή την ε, μαύρη λίστα. Στη μελέτη μας λοιπόν ε, στο 2012 πήραμε τα στοιχεία από το Μνημόνιο των Παρισίων και την ε, Αμερικανική εκτοφυλακή και έχουμε σε αυτό το μήνακα που βλέπετε τα 15 κράτη που προσφέρουν αυτή τη σημαία ευκαιρίας στα πλοία κατηγορίας 1 και μας βλέπουμε πόσες φορές εμφανίζονται τα κράτη 7 στο πίνακα αυτό από τότε που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά η λίστα από το 2000 και μετά. Τα 15 βασικά ε, κράτη εμφανίζονται ξανά και ξανά και είναι στο στόχαστρο της μαύρης λίστας της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και του Μνημονίου των Παρισίων. Και ε, εξαιρέσεις είναι το Ιράν, η Συρία και η Βόρεια Κορέα γιατί τα πλοία που έχουν αυτές τις σημαίες δεν επιτρέπεται να ε, προσαράξουν, να ελιμενιστούν μάλλον στα, στους Αμερικανικούς λιμένες. Με την εξαίρεση της Λιβερίας και της Κίνας, θα έλεγα ότι εκεί έχουμε τις χειρότερες επιδόσεις. Θέλω όμως να σχολιάσω το θέμα της Κύπρου και να πω ότι τα στοιχεία τους έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Ε, η σημαία Κύπρου δεν βρίσκεται στη λίστα του Μνημονίου του Παρισίων εδώ και αρκετά χρόνια τώρα. Γιατί μιλούμε λοιπόν. Λυπούμε για ένα σύνδεσμο ε, που θα βασίζεται στην ποιοτική ανάλυση. Με τη βάση δεδομένων VMIT, το 87% των πλοίων που μπαίνουν στην κατηγορία 1 έχουν ένα μητρό ελέγχων και επιθεωρήσεων πάρα πολύ φτωχό, επιδόσεις φτωχές από πλευράς λιμένων, αν υπάρχουν κιόλα. Επομένως, τίνουν αυτά τα πλοία να κάνουν τις περισσότερες συγκρούσεις, να έχουν τα περισσότερα συμβάντα ρήπανσης ή μόλυσης και να ε, παρουσιάζουν συμβάντα διαρθρωτικής, ε, ε, αν θέλετε, ανεπάρκειας. Και παρόλο που δεν μπορέσαμε να κάνουμε εμπειρική μελέτη αυτή τη στιγμή, οι δείκτες υποδεικνύουν ότι θα μπορούσαμε αυτό το πλέγμα να το εφαρμόσουμε και σε άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη διάπραξη δικημάτων κατά την αυσιπλοεία, όπως είναι η λαθρέα παράνομη αναρχή αλληλεία, η παράνομη εναπόθεση τοξικών αποβλήτων στην θάλασσα και πειρατεία βεβαίως σε ορισμένες περιπτώσεις. Και αν έχω χρόνο θα ήθελα να σας ευχηθήσω την προσοχή και σε άλλα ευρήματα της ε, μελέτης. Όμως νομίζω ότι ε, είπα αρκετά για τη συζήτηση σήμερα. Διάβασα την εξαιρετική έκθεση της συναδέλφου Άννα Γκόμες και των συναδέλφων της. Θεωρώ ότι πράγματι μπαίνει, ε, ασχολείται με το πυρήνα των ζητημάτων, έτσι το αντιλαμβανόμαστε και εμείς, χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου θα πρέπει να εξοικονομηθούν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία, τους μηχανισμούς, ε, τις δυνατότητες που έχει ήδη αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε ευρύτερους στόχους που έχουμε ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να πετύχουμε. Και είναι βασικό αυτό το οποίο ονομάζουμε Safety Security Nexus. Ε, αυτό είναι πραγματικότητα, είναι γεγονός δηλαδή πλοία που εμπλέκονται στο έγκλημα και σε παράνομη δραστηριότητα, λαθρεμπόριο βασικών αγορών, έχουν και πολύ χαμηλά στάνταρ ασφάλειας και θα πρέπει να παρακολουθούνται ε, στενά. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια βιώσιμη και ολιστική προσέγγιση. Είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε. Η έκθεση το τονίζει διότι αυτές οι προκλήσεις είναι διεθνικές, εξού και πολύ περίπλοκες. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουμε να εξοικονομήσουμε κονδύλια και για να το κάνουμε αυτό θα συγκεντρώσουμε όλους αυτούς τους πόρους και τους μηχανισμούς για να έχουμε εξοικονόμηση. Ε, μας έδειξε ε, η ρύθμιση αυτή για την, ε, μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας για την αποκοινού χρήση αεροπλανοφόρων μας έδειξε ότι το ευρωπαϊκό ναυτικό εν γέννη βαίνει συρρυκνούμενο. και αυτή τη στιγμή γίνονται περικοπές στον τομέα της άμυνας και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία στο επίκεντρο οποιασδήποτε στρατηγικής για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας θα πρέπει να είναι η ασφάλεια των ανθρώπων, η σωστή ε, διαχείριση, διακυβέρνηση και ανάπτυξη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία στις ε, δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε το οικονομικό ε, κόστος, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το μεγάλο ατύχημα, το Deep Water, Horizon που έλαβε χώρα το 2010. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αναμορφωθεί η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, ε, βρίσκοντας τους διαφόρους συνδέσμους και ορίζοντας συγκεκριμένους κοινού στόχους, ε, κινδύνους έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και αυτό το προσχέδιο έκθεσης που για μας είναι ύψης της σημασίας. Άρα, συνοψίζοντας, δεν μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε, δεν ενδιαφέρει μόνο να γνωρίζουμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μία πραγματογνωμοσύνη σε σχέση με τις ικανότητες για να δημιουργηθεί μία ε, στρατηγική, ευρωπαϊκή στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας και μόνον. Για μας έχει σημασία κατά πόσο υπάρχει η πολιτική θέληση έτσι ώστε να αρθεί η γραφειοκρατία και να φτάσουμε σε κάτι τελειότερο. Γι' αυτό πιστεύω ότι η συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και περνάμε στο δεύτερο ομιλητή, στον κύριο Διέγκο Εκούνια. Έχετε το λόγο. Thank you uh, for Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι με καλέσατε να ασχοληθώ με αυτό το θέμα ως προς την ε, θαλάσσια διάσταση ασφάλειας της ΚΕΠΑ. Θα ήθελα να πω ότι το έγγραφο αυτό είναι ιδιαίτερα επενεταίο γιατί ασχολείται με θέματα ασφάλειας, ορίζει τις απειλές και μιλά για ολιστική προσέγγιση και συντονισμένη προσέγγιση μέσω μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη θαλάσσια ασφάλεια με ενδιαφέρει η προστασία των ε, θαλασσίων συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό μιλάμε και για εκπόνηση μιας νέας στρατηγικής. Το σημείο εκκίνησης είναι να ε, δούμε τη θεμελιώδη θαλάσσια διάσταση η διάσταση ναυσιπλοείας στις βασικές ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η παγκοσμιοποίηση αφορά το εμπόριο πρωτίστως. Το εμπόριο είναι το διεθνές ε, εμπόριο μέσω θαλασσίων οδών, θαλάσσιας μεταφοράς. Αυτό σημαίνει επιμελητιακή υποστήριξη, ε, ελιμανισμό, μεγαλύτερα πλοία, καθαρά πλοία και βεβαίως και την ε, ναυπηγική καθεαυτή. Αυτά αποτελούν την παγκοσμιοποίηση. Μία άλλη πρόκληση είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Ο εφοδιασμός ενέργειας, μιλάμε για ορυκτά, μιλάμε για ε, υπεράκτιες γεωτρήσεις και για το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να εξαρτώμεθα από μεταφορές μέσω αγωγών, αλλά καλύτερα μέσω θαλασσίων μεταφορών, μέσω τάνκερ. Αυτό είναι και ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε επίσης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που λαμβάνουμε ε, από ε, την ανοιχτή θάλασσα. Αφορά την αιωλική, στη Βόρειο Θάλασσα και ούτω καθεξής. Όταν μιλάμε για τις κλιματικές αλλαγές δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον ρόλο των ε, ωκεανών μέσα στα πλαίσια του ελέγχου και της ε, πόντισης αλλά και της αποθήκευσης ενεργειακών πηγών. Μας ενδιαφέρει ένα κλιματικό πρότυπο και μία προσαρμογή, προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, ε, θέματα ε, αύξησης της στάθμης της θάλασσας και αλλαγές στις ε, παράκτιες περιοχές της Ευρώπης. Πόσο συχνά συνδέουμε τις κλιματικές αλλαγές με τους ωκεανούς. Δυστυχώς πολύ σπάνια. Επίσης χάνουμε σε βιοπικιλότητα Και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταματήσει αυτή την απώλεια της βιοπικιλότητας. Το 80% της ζωής αφορά τη ζωή στους ωκεανούς. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ε, βιωσιμότητα των ωκεανών. Και τέλος, η ασφάλεια καθεαυτή. Έχουμε ταχεία αύξηση απειλών, μη συμβατικών απειλών και στον τομέα των θαλασσών. Κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Αν δούμε αυτές τις προκλήσεις και τις συνδυάσουμε με την Ευρώπη, τότε αυξάνεται η διάσταση του, της θαλάσσιας, των θαλάσσιων μεταφορών γιατί η Ευρώπη είναι μια μεγάλη θαλάσσια υπερδύναμη, η μεγαλύτερη θαλάσσια υπερδύναμη στον κόσμο. Η Ευρώπη ελέγχει το 40% του παγκοσμίου εμπορικού ναυτικού. Έχει 1.200, ε, 1.200 λιμένες και είναι η πρώτη περιφέρεια στην, στις γεωτρήσεις και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στον ε, θαλάσσιο τουρισμό. Έχουμε το μεγαλύτερο ε, τζίρο στη ναυπηγική. Όχι σε τον βεβαίως. Και έχουμε και τον μεγαλύτερο παγκόσμιο εξοπλισμό. Υπάρχει ε, τεχνολογία, υψηλή τεχνολογία θαλασσών Όλα αυτά μας δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο συμφέρον ως προς το θαλάσσιο αυτό ορίζοντα της Ευρώπης. Μιλάμε για ηγετική θέση της Ευρώπης και αυτό για τη γεωγραφική της θέση πρωτίστως. Έχει την μεγαλύτερη γραμμή παρακτήων περισσότερο από τη Ρωσία ή άλλες ε, περιοχές του κόσμου και από την Ασία. Είναι μια μεγάλη χερσόνησος η οποία ε, πλαισιώνεται από νησιά και γι' αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, ότι προωθούμε την αυσυπλοεία. Έχουμε τέσσερις χώρες οι οποίες είναι νησιά και υπάρχουν η Ελλάδα, η Δανία, η Ισπανία και η Πορτογαλία και η Ιταλία που είναι χερσόνηση. Αυτό μας διανοίγει οδούς προς άλλες αγορές. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι υπάρχει θαλάσσια διάσταση, αυτή η θαλάσσια διάσταση στην ασφάλεια στην ΚΕΠΑ της Ευρώπης και μιλάμε για ελεύθερο εμπόριο, το οποίο σημαίνει ελευθερία ναυσιπλοείας πρωτίστως. Χρειάζεται λοιπόν παγκόσμια ασφάλεια στους ωκεανούς. Αυτό ε, αφορά τις ε, θαλάσσιες οδούς και τη ε, ναυσιπλοεία τους. Υπάρχουν θαλάσσια συμφέροντα τα οποία ε, άπτονται των οικονομικών, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ειρήνη στους ωκεανούς για να προωθηθεί αυτό το εμπόριο. Μιλάμε για βιωσιμότητα των ωκεανών που έχει μεγάλη σημασία να είναι ασφαλής η ωκεανοί μας για τις παράκτιες περιοχές το 40% του πληθυσμού της Ευρώπης ε, ε, ζει σε παράκτιες περιοχές και το 50% του ΑΕΠ παράγεται σε παράκτιες περιοχές. Γι' αυτό και η αλληλεία είναι ύψης της σημασίας στην Ευρώπη, στην Ευρώπη και αλλού. Όχι μόνο λόγω των αλλιευτικών αποθεμάτων, αλλά και εκ του γεγονότος ότι είμαστε και οι μεγαλύτεροι καταναλωτές στην Ευρώπη. Μιλάμε για 30% ανακεφαλή κατέτος, ενώ αλλού είναι κάτω από, 20 κιλά ανακεφαλή και αναέτος. Η βιωσιμότητα έχει σημασία και για τον τουρισμό αναψυχής και το 66% ε, των τουριστικών δραστηριοτήτων αφορά ε, δραστηριότητες αναψυχής με βάση την αυσιπλοεία. Αυτό αφορά και το περιβάλλον στη συνέχεια. Ως προς τις ε, κλιματικές αλλαγές αποτελούν απειλή μακροχρόνια, πολύ περισσότερο από άλλες συμβατικές απειλές. Η γεωργία η αλληλεία ορίζονται από τους ωκεανούς, γι' αυτό η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η διάβρωση των ακτών, όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία για τις ε, παράκτιες ε, περιοχές. Και θα πρέπει να δούμε πώς οι κλιματικές αλλαγές ε, επιδρούν στις αλλαγές του θαλασσίου ορίζοντα το 40% του πετρελαίου και το 60% του φυσικού αερίου ε, λαμβάνονται από ε, γεωτρήσεις τους ανοικτούς ωκεανούς. Γι' αυτό μίλησα για την αυτονομία μας από τους αγωγούς μεταφοράς ε, φυσικού αερίου και πετρελαίου. Γι' αυτό η γεώτρηση αποτελεί μια τάση η οποία αναπτύσσεται, όλο ένα και περισσότερο. τα αεολικά πάρκα η βιομάζα, τα βιοκαύσιμα, όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία γιατί σχετίζονται άμεσα με τους ωκεανούς και τις θάλασσες. Γι' αυτό και η ενέργεια άπτεται των θαλασσίων συμφερόντων της Ευρώπης. Ως προς την ασφάλεια σε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες, η ασφάλεια είναι ύψης της σημασίας για τις θαλάσσιες οδούς της Ευρώπης. Της Και οι συνάδελφοί μου ασχολήθηκαν και θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Τα δύο τρίτα των συνόρων είναι παράκτια ε, σύνορα στην Ευρώπη και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτή την ε, διάσταση της ασφάλειας στην ΚΕΠΑ. Δεν μιλάμε παρά για συγκεκριμένες απειλές. Μιλάμε για παράνομη μετανάστευση, λαθρεμπόριο, δουλεμπόριο, απειλές οι οποίες ολοένα και διονγκούνται στην ε, Αρκτική, στη Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα. Μπορούμε να πούμε ότι σε δύσκολους καιρούς και καιρούς κρίσης που διανύουμε, αυτό είναι αναπόφευκτο και γι' αυτό ίσως η θαλάσσια ασφάλεια είναι ίσονο σημασίας. Ισχύει όμως ακριβώς το αντίθετο. Σε τέτοιο καιρό κρίσης ξεκινάμε από το μηδέν, δηλαδή λαμβάνουμε υπόψη τις γεωγραφικές μας βάσεις και στη, μιλάμε για τη βιώσιμη χρήση των ε, ε, θαλασσών μας γιατί η θάλασσα και οι ωκεανοί επέτρεψαν την συσσόρευση κεφαλαίου στους λαούς μας. Και όταν σκεφτόμαστε, μιλάμε για την Ευρώπη, λαμβάνουμε υπόψη την αυσιπλοεία. Αρχίσαμε με τους Βίκινγκς, τους θαλασσοπόρους, τους Ήβυρες και ούτω καθεξής. Δεν μιλάμε μόνο για τη γεωγραφία μας, αλλά και για την κοινή μας ιστορία. Όταν μιλάμε για ε, πολιτικές ε, πλαίσιο σε σχέση με τα θαλάσσια συμφέροντα, μιλάμε για τη θαλάσσια πολιτική μας, που είναι ένα πολύ βασικό βήμα, διότι για πρώτη φορά οι Βρυξέλλες αντιμετώπισαν τις θάλασσες ολιστικά λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εμπλεκόμενες πτυχές. Μία νέα στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας αποτελεί τον χαμένο κρίκο, τον οποίο βρήκαμε. Αρχικά η Κομισιόν ασχολήθηκε με το θέμα, αλλά η Κομισιόν έχει πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες τομείς της ΚΕΠΑ. Γι' αυτό μιλήσαμε και για ασφάλεια, αλλά και για εποπτεία των θαλασσών στην Ευρώπη. προωθήσαμε και μία περιβαλλοντική πολιτική μέσα στα πλαίσια της θαλάσσιας πολιτικής ασφαλείας Πρόκειται για μια ειδική οδηγία πλαίσιο για την θαλάσσια ασφάλεια και με βάση την ε, θαλάσσια έρευνα και υπάρχει και μια οδηγία για τη θαλάσσια έρευνα. Και λάβαμε υπόψη και την εδαφική διάσταση των ε, θαλασσίων οδών ήδη την προηγούμενη εβδομάδα με βάση την προτινόμενη οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά υπάρχει και αυτός ο χαμένος κρίκος, όπως σας είπα, ως προς την ασφάλεια. Είχαμε τα ατυχήματα του Εύρικα και αρχικά και του Πρεστής και δεν μπορέσαμε να βελτιώσουμε την διάσταση της ασφάλειας. Αν δείτε την Μεσόγειο, Βλέπετε ότι υπάρχει μια κατάσταση status quo. Δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι μια στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας για την Ευρώπη δεν θα πρέπει να αποτελέσει επικάλυψη της ε, θαλάσσιας πολιτικής. Τα θαλάσσια συμφέροντά μας ως προς την ασφάλεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με συμφέροντα ενέργειας κλιματικών και κλιματικών αλλαγών. Αλλά δεν θα πρέπει να προωθούμε επιμέρους ολοκληρωμένες πολιτικές που έχουν καλυφθεί από θέματα θαλάσσιας ασφάλειας. Μιλάμε για μία πολιτική που εστιάζεται στην ασφάλεια, στην εποπτεία, στρικτοσένσου, αλλά δεν ε, προβαίνουμε σε επικαλύψεις ως προς την εργασία που έχει γίνει το τελευταίο καιρό στον τομέα της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της έρευνας. Μιλάμε για μια πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας ε, στις θάλασσες, και όταν μιλάμε για την Ευρώπη, μιλάμε για μια ήπειρο που είναι τρεις φορές μικρότερη από την Αφρική ως προς μάζα ε, γης, αλλά η ε, ακτογραμμή της είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη της Αφρικής. Γι αυτό Γιατί θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε μία θαλάσσια πολιτική ασφάλειας. Ε, για λόγους γεωγραφίας, μα γιατί άλλο βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Και τέλος, ο αντινάφαρος κύριος Φέλτ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ευρωβουλευτές, κυρίε και κύριοι, τα επόμενα 12 με 15 λεπτά θα περιγράψω πολύ σύντομα ορισμένες πλευρές του τομέα της ναυσιπλοείας που έχουν ε, επιπτώσεις στην κοινή πολιτική ασφάλειας άμυνας και θα κάνω ε, διατύπωση πορισμάτων στο τέλος. Δεν θα μπορέσω να τα καλύψω όλα βέβαια, αλλά προσβλέπω και στις ε, ερωταπαντήσεις η ενίσχυση της ε, ανασφάλειας ε, στις θάλασσες λόγω της τρομοκρατίας, της παράνομης μετανάλευσης και των ασυμμετρικών απειλών που προκαλούνται από ε, εγκληματίες και κυβερνήσεις καταδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη ασφάλεια, ενεργή, παθητική και άμυνα στον τομέα της θάλασσας. Πρέπει να υπάρχει πιο συντονισμένη συλλογική δράση για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πολύ διαφορετικές προκλήσεις. Πολλές χρήσιμες πρωτοβουλίες ήδη διεξάγονται υπό την αιγίδα και των κρατών μελών και της ίδιας της Ένωσης. Η πολιτική για την ενιαία ε, πολιτική για τις θάλασσες και την αυσιπλοεία της Κομισιόν και το σχετικό πρόγραμμα για ένα κοινό περιβάλλον ε, ε, διανομής πληροφοριών είναι ενθαρρυντικές εξελίξεις. Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες που ήδη λειτουργούν καλά, όπως το ΡΙΚΑΠ στην Νοτιοανατολική Ασία, και το ε, σύστημα για την ε, αναγνώριση των στόχων ραντάρ και το θαλάσσιο σύστημα ασφάλειας ενεργητικής και παθητικής ε, είναι συστήματα που λειτουργούν με όλα τα 65 κράτη-μέλη. Είναι ε, συστήματα που προσπαθούν να καταπολεμήσουν τους συνολικούς, τις συνολικές αυτές απειλές. Προσπαθούν να ενισχύσουν την ασφάλεια και την άμυνα στον τομέα της ναυσιπλοείας. Ο πρώτος στόχος είναι η ε, κοινή χρήση των πληροφοριών. Πρέπει να περάσουμε από ε, την αντιμετώπιση της ε, διανομής της πληροφόρησης με βάση την ανάγκη γνώσης, στην διανομή της πληροφόρησης με βάση την αρχή της ευθύνης για την διανομή των πληροφοριών. Υπάρχουν πολλά που ξέρουμε, πολλά που δεν ξέρουμε, αλλά το πιο κρίσιμο είναι αυτά που δεν ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε. Γιατί υπάρχουν πράγματα που ξέρουμε ότι ξέρουμε και πράγματα που ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε. Για τον τομέα της ε, ενεργητικής και παθική ασφάλειας ε, στις θάλασσες είναι πολύ βασικό. Οι αρχές αυτές είναι η βάση της ασφάλειας των θαλασσών. Η αρχή της διανομή ε, πληροφόρηση διανομής με βάση το ποιο πρέπει να τη γνωρίζει είναι μια απαρχαιωμένη αντιμετώπιση τότε που η πληροφόρηση διανεμόταν ε, μέσω ορισμένων ε, ε, και πολύ συγκεκριμένων και περιορισμένων συχνοτήτων, που ήταν βεβαίως πολύ περιορισμένα δίκτυα. Αντίθετα σήμερα, η ζωή των, και των μηχανών και των λογισμικών είναι πολύ μικρή και όλη η πληροφόρηση μπορεί να ληφθεί από το ίντερνετ και διάφορα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Θέλουμε λοιπόν μια αλλαγή στην οτροπία να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα για την ε, κοινή χρήση των πληροφοριών στον τομέα των θαλασσών. Θαυμάσιο παράδειγμα έχουμε στον τομέα των αεροπορικών συγκοινωνιών, όπου υπάρχει ανοιχτή ανταλλαγή πληροφοριών εδώ και πολλά χρόνια και που συνεχώς βελτιώνεται. Η δεύτερη αρχή είναι η επιτήρηση των θαλασσών, που να μας δίνει μια εικόνα για την κατάσταση στη θάλασσα για όλους όσους συμμετέχουν στην δραστηριότητα στον τομέα αυτό έχουμε ευθύνη σε τρία επίπεδα. Στρατηγική ευθύνη, λειτουργική ευθύνη και τακτική ευθύνη. Αλλά ποιοι είναι οι κύριοι φορείς που ασχολούνται σε συνολικό και περιφερειακό τομέα. Το αντίθετο της ε, συνειδητοποίησης της ανάγκης ε, πληροφοριών για τη θάλασσα είναι η τυφλότητα στις θάλασσες. Υπάρχουν διάφοροι φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη-μέλη ή θεσμικά όργανα που δεν καταλαβαίνουν την ανάγκη για πληροφόρηση στον τομέα της θάλασσας, κάτι που υπάρχει και σε εθνικά κοινοβούλια και σε κοινοτικές αρχές. Χρειάζεται ρωμαλαία ασφάλεια στον τομέα των θαλασσών. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε τη σημασία της θάλασσας για την ευημερία και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μέσω των θαλασσών ε, γίνεται εμπόριο, είναι πηγή για τροφή, είναι πηγή για ενέργεια, και χρειαζόμαστε λοιπόν καλή διακυβέρνηση. Για πολλούς όμως η θάλασσα είναι και ο φορέας για παράνομες, επικίνδυνες και εγκληματικές δραστηριότητες. Εάν δεν αναγνωρίσουμε πλήρως αυτή την κατάσταση, εάν δεν αλλάξει η πολιτική όπως πρέπει, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη ανάγκη για ασφάλεια των θαλασσών ικανοποιητικά. Υπάρχουν έξι στρατηγικοί φορείς που ασχολούνται με την ασφάλεια και άμυνα στον τομέα των θαλασσών. Ο πρώτο είναι τα Ηνωμένα Έθνη μέσω του Διεθνού Οργανισμού Ναυσιπλοεία. Ο δεύτερο είναι οι ακτοφυλακοί, οι πεζοναύτε και το ναυτικό των Ηνωμένων Εθνών μέσω τη κοινή στρατηγική και η κυβέρνηση μέσω τη υποστήριξη που δίνει στο Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοεία. Ο δεύτερο είναι το ΝΑΤΟ, γιατί πολλά ναυτικά του κόσμου συμμετέχουν σε αυτόν και υπάρχει και η πολιτική του για την ασφάλεια, ε, για την στρατηγική για την ε, θάλασσα, που λέγεται MSO. Και τέταρτος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Επιτροπής. Η πέμπτη είναι η Αφρικανική Ένωση, ο πέμπτος φορέας, μέσω της πολύ σοβαρής φιλοδοξίας να εφαρμόσει τη δική του στρατηγική για την ασφάλεια των θαλασσών. Και το έκτο είναι αδέσμευτα κράτη όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα, καθώς και το Πακιστάν και η Τουρκία, που προς το παρόν μεμονωμένα έχουν το δικό τους ναυτικό και τις δικές τους ε, φιλοδοξίες και στρατηγικές στον τομέα των θαλασσών. Ω τμήμα των ΗΕ, ο, οργανισμός για την, ε, ο Διεθνής ε, Οργανισμός IMO, υποστηρίζει τις περιφερειακές δραστηριότητες και τις βοηθάει να έχουν αποτελέσματα. Αλλά τα Ηνωμένα έχουν περιορισμένη εμπειρία στον τομέα των θαλασσών και δεν έχουν εντολή να εφαρμόσουν τους ισχύοντες νόμους η πρώτη ε, ναυτική αποστολή των ΗΠΑ είναι το UNIFIL που εφαρμόζει το εμπάργκο όπλων εκτός των ακτών του Λιβάνου. Τα Ηνωμένα Έθνη δρούν σε τρία επίπεδα και σε στρατηγικό και σε λειτουργικό και τακτικό και υποστηρίζουν τον IMO μέσω του, της, ε, ε, εάν, παρά το ότι η γερουσία των ΗΠΑ δεν έχει εφαρμόσει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Η ταχεία, η ταχεία εφαρμογή των ε, κωδικών για την ασφάλεια μετά τις επιθέσεις της 9 ε, Σεπτεμβρίου αποδεικνύουν την πολιτική βούληση των ΗΕ. Το ΝΑΤΟ έχει οθετήσει και την στρατηγική ασφάλεια και την αρχή για την ασφάλεια στον τομέα της θαλάσσης. Η στρατηγική για τις θάλασσε ε, πέρα από καθαρά στρατηγική, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ έχει γίνει πιο σφαιρική, συνδέοντας και πολιτική και στρατηγική πλευρά και δίνει υψηλότερη προτεραιότητα στην ε, στρατηγική για την ασφάλεια των θαλασσών. Το ΝΑΤΟ θέλει να δράσει σε όλα τα επίπεδα, ανάλογα με την πολιτική βούληση των κρατών που το αποτελούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλεια με τρει στόχου. Να αντιμετωπιστεί η πρόκληση, να οικοδομηθεί η ασφάλεια στην περιοχή και να επιτευχθεί μια διεθνή τάξη που να βασίζεται σε αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση. Αυτή η στρατηγική προπήρχε τη συνθήκη τη Λισαβόνα η οποία συνθήκη τη Λισαβόνα καλεί για περισσότερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ευρωπαϊκών οργανισμών και τρίτων χωρών. Ένα ρόλο των συλλογικών υπηρεσιών θα ήταν να βοηθήσουν τη διαδικασία συντονισμού και συνεργασία για μερικά θαλάσσια καθήκοντα, τα άρθρα 47 και 222 τη συνθήκη τη Λισαβόνα δίνουν καθαρή καθοδήγηση για το πώ πρέπει να δράσουμε για να προλάβουμε τρομοκρατική απειλή στην επικράτεια των κρατών μελών. Η Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητε και στρατιωτικές που παρέχουν τα κράτη-μέλη. Το άρθρο 222 της συνθήκης αναφέρει επίσης τις ε, θεομηνίες ε, ή, τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να είναι βάση για να ζητηθεί από τα κράτη-μέλη βοήθεια. Θα μπορούσε να έχει μια μόνιμη ε, ναυτική δύναμη όπως η Euromar Force στην Μεσόγειο και η Επιχειρήσει του Frontex στη Μεσόγειο είναι σημαντικό τμήμα για να επιτευχθεί καλή κατάσταση στη θάλασσα. Για παράδειγμα, η Αταλάντα μαζί με, τη, με το πρόγραμμα για τη δημιουργία ε, θαλάσσιας ε, δυνατότητας ε, στον, στο κέρας της Αφρικής θα ήταν ένα μεγάλο βήμα για περισσότερη συνεργασία από πλευράς Κομισιών. Ποιες τώρα είναι οι απειλές, τα ευάλωτα σημεία και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Ένωση και ο πληθυσμός της έχουμε τρία κεφάλαια. Το πρώτο είναι οι απειλές που αφορούν άμεσα την επικράτεια και τους πολίτες από τη θάλασσα. Το δεύτερο, οι απειλές που αφορούν τα σφαιρικά θαλάσσια συμφέροντα και το τρίτο είναι οι απειλές που, ε, κατά των πόρων που βρίσκονται στη θάλασσα. Και οι τρεις, τομείς και και αυτοί τομείς αφορούν απειλές που μπορείτε να βρείτε και στο σχέδιο έκθεσης που σας έδωσα. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συνέστηση ότι οι απειλές αυτές είναι σφαιρικές. Άρα και οι απαντήσεις μας πρέπει να είναι σφαιρικές. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι και άλλες ε, εγκληματικές και παράνομες δραστηριότητες στη θάλασσα δεν επηρεάζουν μόνο την Ευρώπη, αλλά και άλλες κράτης, άλλα κράτη παντού στον πλανήτη. Για παράδειγμα, η λαθρομετανάστευση και το λαθρομπόριο ναρκωτικών μέσω των θαλασσών αποτελούν σημαντικές εσωτερικές απειλές για την Ένωση. Ήδη αναφέρθηκα στην παράνομη, ανεξέλεγκτη και άναρχη ε, αλληλεία, την απόρριψη τοξικών ουσιών, την παράνομη τροφοδότηση σε καύσιμα. Όλα αυτά ε, υπονομεύουν την οικονομική βιωσιμότητα των κρατών μελών. Ορισμένα αδύνατα ή καταργημένα κράτη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτέ τι απειλέ. Αυτό συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση. Μια, ένα άλλο ευάλωτο σημείο προκύπτει από το μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων που ε, ζουν και εργάζονται εκτό Ευρώπη ή δουλεύουν σε διάφορε επιχειρήσει ε, εκτό Ευρώπη ή εργάζονται ω μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων. Επίση οι τουρίστες είναι επίση τρωτοί γιατί όλο και πιο συχνά προσελκύονται από διάφορους συναρπαστικούς και εξωτικούς ε, τουριστικούς προορισμούς, ανεξάρτητα από τους κινδύνους. Πολλές φορές χρειάστηκε να γίνουν ε, επίγουσες ε, εκενώσεις πληθυσμών Οι πολιτών μας και διάφορα κράτη-μέλη βοήθησαν για να εξαχθούν πολλοί πολίτες είτε με ίδια πρωτοβουλία είτε μετά από συστάσεις από τοπικές αρχές. Ορισμένοι έχουν μια μόνιμη ναυτική παρουσία σε, κάποιους, ε, σε κάποιες περιοχές όπου υπάρχουν συγκρούσεις όπως ο κόλπος της Γουινέας για να μπορέσουν να παρέμβουν σύντομα. Η ρήτρα αλληλεγγύης στη συνθήκη της Λισαβόνας δεσμεύει τη Λισαβόνα μέσω της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης να έχουν πιο μόνιμες ρυθμίσεις. Καταλήγοντας, είναι σαφές ότι η στρατηγική μας στον τομέα αυτό είναι αναγκαία, που να βασίζεται σε μερικές αρχές. Δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί πόσο δύσκολο θα είναι να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, αλλά πόσο θα βελτιώσει την κατάσταση. Οι αρχές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συλλογική και μόνιμη πολιτική βούληση, ηγεσία και δέσμευση. Και επαναλαμβάνω, χρειάζεται συλλογική και μόνιμη βούληση, ηγεσία και δέσμευση. Και αξιόπιστη δυνατότητα παρέμβαση οποιοδήποτε μείγμα πολιτική και στρατιωτική δύναμη. Μια ολιστική, σφαιρική προσέγγιση για όλα τα θέματα ασφάλεια που έχουν θαλάσσια διάσταση. Να καταλάβουμε ότι το θαλάσσιο πλαίσιο είναι παγκόσμιο, άρα και οι απαντήσει πρέπει να είναι παγκόσμιες. Να έχουμε μια περιφερειακή και όχι συγκεντρωτική προσέγγιση. Να ενθαρρύνουμε εξελικτικά βήματα, όχι ριζικά. Να επιδιώξουμε να επιβάλλουμε όρια στη θάλασσα, να διαχωρίσουμε τα όρια των επιχειρήσεών μας μεταξύ των κρατών μελών είναι απλώς αντανάκλαση μιας παροχημένης αντίληψης και δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε δράσης. Όλα τα κράτη-μέλη που έχουν αρχές για επιβολή του δικαίου της θάλασσας θα πρέπει να κάνουν ασκήσεις για συλλογικές δράσεις, ούτω ώστε οι διαφορετικές δυνατότητες και περιορισμοί τους να γίνουν κατανοητοί και να ληφθούν υπόψη. Πρέπει να επεκτείνουμε την σταθερότητα από την Ευρώπη προς τα έξω. Αυτό χρειάζεται ένα όραμα, πολιτική βούληση, γενοδορία και παρατεταμένη δέσμευση. Η πολιτική προτεραιότητα είναι το σύνεκ βανών. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έχει τα αναγκαία μέσα για να παίξει το ρόλο της, για να εγγυηθεί τα συμφέροντα των πολιτών της. Η συνθήκη της Λισαβόνας επιτρέπει την ε, αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των, των, των ε, πυλώνων όπως αποκαλούσαμε προηγουμένως, αλλά αυτό θέλει θάρρος. Συνεχή πολιτική βούληση και στήριξη. Καταλήγοντας, η, η κύρια σύστασή μου είναι να αναπτύξουμε την περιφερειακή διάσταση όλων των δραστηριοτήτων μας που σχετίζονται με την ασφάλεια των θαλασσών σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές που είναι γύρω από την Ευρώπη. Πρέπει να ε, συμμετάσχουν και συνεργαστούν όλοι οι φορείς με σαφή και ισότιμη ε, κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων, όπως είναι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα πολιτικά επιτελεία. Για να το επιτύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε επιγόντω μία στρατηγική για την ασφάλεια των θαλασσών. Με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρος. Θα έπρεπε να ε, μιλάτε λίγο πιο αργά, λέει ο Πρόεδρος. Με συγχωρείτε, αλλά μια πρόταση έχω. Μια πρόταση την οποία θα διαβάσω πολύ αργά. Για να το επιτύχουμε χρειαζόμαστε επιγόντω μια τέτοια λοιπόν στρατηγική, ευρωπαϊκή στρατηγική που θα αναπτυχθεί από κοινού με όλες τις ε, αρμόδιες αρχές. Πρέπει να αποκλείσουμε, εάν συνειδητό αποκλείσουμε οποιαδήποτε αρχή από αυτήν την ε, διαδικασία, θα υπονομεύσουμε την επίπτωση αυτή της στρατηγικής. Γι' αυτό Χρειαζόμαστε ισχυρή πολιτική βούληση και ηγεσία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές για την παρέμβασή σας, αλλά και για το ότι τηρήσατε ε, την, ε, το χρονικό όριο που είχατε. Ποιος από τα μέλη θέλει να θέσει ερωτήσεις. Πρώτα ο κύριος Γκάλερ. Να πω στα μέλη, στους βουλευτές, ότι καλό θα είναι να μην ξεπεράσουν τα τρία λεπτά ο καθένας στην παρέμβασή του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Νομίζω ότι και οι τρεις ήταν ε, πολύ χρήσιμες. Αυθόρμητα θα μπορούσα να συμφωνήσω με όλα όσα υπόθηκαν ως ανάλυση και με τα πολιτικά πορίσματα που εξήχθησαν. Είναι νομίζω σαφές ότι υπάρχει πολιτική βούληση για όλα αυτά που θέλουμε. Όλοι το ανέφεραν. Όχι, χρειαζόμαστε να υπάρχει πολιτική βούληση καλύτερα. Και γι' αυτό καθήκον και της δικής μας υποεπιτροπής είναι να λάβουμε την πρωτοβουλία να γίνουν αυτές οι ενέργειες για να υπάρξει αυτή η πολιτική βούληση και στην Ολομέλεια και στα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ότι η κατάσταση τη συνθήκη τώρα καθιστά δυσχερές να χρηματοδοτηθούν μέτρα στον τομέα ασφάλειας και άμυνας. Γιατί εδώ χρειαζόμαστε άμεσα τα κράτη-μέλη. Εφόσον λοιπόν επιδιώκουμε μια στρατηγική για την θαλάσσια ασφάλεια και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, έχουμε όλοι το ίδιο συμφέρον και υφιστάμεθα όλοι τις ίδιες απειλές. Ξέρουμε ότι η ναυσιπλοεία όλων των κρατών μελών, μελών μας από εδώ μέχρι την Ανατολική Ασία περνάει από τα ίδια δρομολόγια. Ξέρουμε επίσης ότι η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου μαζί με τους εταίρους μας πρέπει να βασιστεί κατόπιν, δηλαδή το προϊόν της εκμετάλλευσης, πρέπει να πάει από τις ίδιες διαδρομές για να επανέλθει στην Ευρώπη. Όμως πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη στον ίδιο βαθμό σε θέση να δράσουν στον τομέα των θαλασσών. Ορισμένοι δεν είναι καθόλου σε θέση. Ορισμένοι δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν την προσπάθεια. Υπάρχουν κράτη που μπορεί να μην έχουν ε, πολύ εκτεταμένες ακτογραμμές, αλλά παρόλα αυτά έχουν ε, εκτεταμένο θαλάσσιο εμπόριο και ενδιαφέρονται. Γι' αυτό, για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας, τα οικονομικά μας συμφέροντα στη θάλασσα, θα έπρεπε πολλά να κάνουμε και πρέπει να διαχωρίσουμε σε ποια ακριβώς μέτρα μπορούμε, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, να συγχρηματοδοτήσουμε προσπάθειες. Εάν, για παράδειγμα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδοτούμε προσπάθειες και σκάφη, αυτό θα σήμαινε να καταλάβουμε ότι όλοι χρησιμοποιούμε τα ίδια δρομολόγια, όλοι έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Οι καιροί όπου διάφορα κράτη-μέλη υποστήριζαν ε, διαφορετικούς πειρατές για να θίξουν κάποια άλλη, άλλα κράτη-μέλη, έχει ευτυχώς, έχουν αυτοί οι καιροί παρέλθει εδώ και κάποιους αιώνες. Οπότε, οι απειλές που υφιστάμεθα μας αφορούν όλους και γι' αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν από κοινού και να συγχρηματοδοτηθούν, τονίζω. Ευχαριστώ κυρία Νικολάη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Συμφωνώ σχεδόν με, με όλα όσα είπατε. Το επόμενο θέατρο διαμαχών θα είναι η θάλασσα, παρόλο που όλοι λένε ότι τους αρέσει η ειρήνη. Και αυτά είναι πράγματα που θα δούμε όλο και περισσότερο να ανακύπτουν τα επόμενα 5, 10 ή 15 χρόνια και δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδου συγκρούσεις. Επομένως, η θαλάσσια διάσταση της πολιτικής ασφάλεια και άμυνας θα αποτελέσει μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την ευρωπαϊκή πολιτική. Έχω κάποια ερωτήματα ω προς την παρουσίασή σα. Είπατε Ε, μιλήσατε για αυτά τα οποία γνωρίζουμε ότι ξέρουμε, για αυτά τα οποία γνωρίζουμε ότι δεν ξέρουμε και για αυτά τα οποία δεν γνωρίζουμε ότι δεν τα γνωρίζουμε. Και γι' αυτό μιλήσατε και για την ανάγκη ε, διάδοσης και διανομής των πληροφοριών. Πιστεύετε ότι από πλευράς διεθνούς δικαίου χρειαζόμαστε νέα προσέγγιση για τη ρύθμιση της θαλάσσιας διάστασης Πρέπει να αξιολογήσουμε και τη σύμβαση αλλά και το θεσμό αν θέλετε το καθεαυτό. Ίσως έχει έρθει η ώρα να αλλάξουμε κάποιο, κάπως, να μπούμε πιο βαθιά στο θέμα. Εσείς τι πιστεύετε. Και από εκεί και πέρα έχουμε αυτό το που αποκαλούμε θαλάσσια γειτονία. η πολιτική μας για τη Μεσόγειο ή για τη Βαλτική θάλασσα δεν έχει ε, τόσο ε, μεγάλη σχέση Interesting uh, thing. με τη Μαύρη Θάλασσα. Και η Τουρκία γίνεται όλο και πιο εμπλεκόμενος παράγοντας στη Μαύρη Θάλασσα και καθώς και η Ρωσία. αλλά και ερχόμενοι στη Μεσόγειο, η οποία δεν έχει σχέση με τη θαλάσσια τόσο διάσταση της Ρωσίας όσο η Μαύρη Θάλασσα. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Δύο μπλόκα έχουμε στη θαλάσσια πολιτική. Το ένα σχετίζεται με την Κίνα, η οποία αναλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην Ασία και τον Ειρηνικό και το άλλο σχετίζεται βεβαίως με τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι ε, μεγάλος παίκτης σίγουρα στον Ατλαντικό και στον Βόρειο Ειρηνικό. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν αυτές οι δύο ε, παγκόσμιες ε, διαστάσεις, αν θέλετε, οι οποίες είναι όλο και πιο παρούσες στη θάλασσα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμα θέλει να μιλήσει τελευταία, γι' αυτό να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Beauty Κόφερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να ομολογήσω ότι έχω Πολλές ερωτήσεις ακόμη. Πρώτα απ' όλα, οι αποτιμήσεις και αναλύσεις του κινδύνου είναι τεκμηριωμένες. Το καταλαβαίνω. Αλλά η σχέση ανάμεσα σε αυτή την τόσο τεκμηριωμένη ε, ανάλυση κινδύνων και τις ε, πραγματικές ε, δυνατότητές μας είναι αμφίβολη. Ο κύριος Γκάλετ είπε ότι θα έπρεπε να συγχρηματοδοτήσουμε ε, σκάφη, πλοία, ένα στόλο δηλαδή. Αλλά κοιτάξτε εδώ είμαστε ανίκανοι να συνεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε από κοινού αυτά που ήδη έχουμε. Οπότε το να έχουμε μια στρατηγική με, τέτοιες, ε, ε, με τέτοια ευχολόγια για μελλοντικά σχέδια δεν νομίζω ότι βοηθάνε να προσανατολιστούμε. Βεβαίως έχουμε εμπορικά συμφέροντα ως Ευρώπη. Τίθεται το ερώτημα εάν στην ε, Νότια Κίνα είναι ασφαλή στην αυσιπλοεία, μας ενδιαφέρει αυτό. Αλλά τι μπορεί να κάνει η κοινή πολιτική ασφάλειας άμυνας σε αυτές τις περιοχές για να υπάρξει περισσότερη ασφάλεια. Θα ήθελα να είμαστε συγκεκριμένοι. Παρακαλώ λοιπόν τους ειδήμονες ποιο είναι το όραμά μας εκτός Ευρώπης. Τι μπορεί να γίνουν τα επόμενα δέκα χρόνια. Τι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Που να έχει έννοια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Και εγώ σας ευχαριστώ, η κυρία Γκόμες. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εμπειρογνώμονες για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους, οι οποίες ε, βασίζονται ε, σε πολύ σημαντικά στοιχεία. Μαθαίνω πολλά από τη δική σας έρευνα και αντλώ στοιχεία από τις μελέτες που εκπονείτε εσείς για τη σύνταξη της δικής μου έκθεσης. Κάτι το οποίο είναι πολύτιμη βοήθεια για εμένα. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τα καλά σας λόγια ως προς την ε, έκθεση τη δική μας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις που προκύπτουν από τις παρουσιάσεις σας. Κύριε Γκρίφιθ. Πώς αξιολογείτε εσείς και το Ινστιτούτο της Στοκχόλμης την πιθανότητα ε, έλευσης κάποιας μεγάλης καταστροφής κάποιες καταστροφές μεγάλου μεγέθους, ε, την οποία να μην μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κράτο, κράτος μέλος από μόνο του και η οποία θα χρειαστεί ε, συντονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο δράση. Για παράδειγμα, όπως η καταστροφή του Horizon Η εξόριξη σε μεγάλα βάθη είναι κάτι στην ανοιχτή θάλασσα που είναι κάτι που εξαπλώνεται όλο και περισσότερο, αλλά και το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων. Υπάρχει επίσης. Συχνά λαμβάνω μηνύματα από πολίτες και μάλιστα από ε, ε, πολίτες ε, της Δανίας από ένα συγκεκριμένο δανό πολίτη που έχει ε, ιστορικό στο ναυτικό, έχει ιστορική διαδρομή στο ναυτικό και ο οποίος συνεχώς μας στέλνει στοιχεία ότι προετοιμάζεται ε, κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο προετοιμάζεται ένα τέτοιο πλήγμα ενδεχομένως εναντίον κάποιας πολύ σημαντικής υποδομής λιμενικής μεταξύ άλλων, κάτι το οποίο θα έχει τεράστιο αντίκτυπο ε, και φοβερές συνέπειες όχι μόνο στην οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, θα έχει και μεγάλο ε, φόρο σε ανθρώπινες ζωές. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που είναι γνωστό ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε σε ευρωπαϊκούς λιμένες προχωρούν σε εποπτεία και ανείχνευση των εμπορευματοκιβωτίων που προορίζονται για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να μην ε, τίθεται υπόψη των Ευρωπαίων πολιτών είναι κάτι για το οποίο προετοιμάζονται οι ευρωπαϊκές αρχές. Από πλευράς ε, ασφάλειας και μόνο. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερον, τι γίνεται εάν προκύψουν συγκρούσεις π.χ. στη θάλασσα της Κίνας, κάτι το οποίο απέφχομαι σφόδρα. Ε, τις συγκρούσεις δηλαδή οι οποίες είναι μακριά από εμάς γεωγραφικά. Μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, μην ασχοληθούμε, να τις παραμελήσουμε και να ασχοληθούμε μόνο με τα άμεσα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. είναι κάτι που είναι απαραίτητο για μια ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θάλασσα ή είναι κάτι το οποίο δεν σχετίζεται με αυτή τη στρατηγική. Αυτές οι δύο ερωτήσεις απευθύνονται στον κύριο Γκρίφιθ. Κύριε Πίτα Ικούνια, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Συμφωνείτε ότι ε, θα ήταν χρήσιμη μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή είναι, είναι μια πρόταση που έρχεται και από άλλες επιτροπές στο Κοινοβούλιο. Στην Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος χθες παρουσιάστηκε το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Γιακολίνο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Και μία από τις προτάσεις είναι η δημιουργία ευρωπαϊκής ακτοφυλακής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κάποια φαινόμενα περιορισμένου μεγέθους οι οποίοι, τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ε, ένα προήμιο για όλα αυτά. Αλλά δεν έχουμε μια ακτοφυλακή ε, ολόκληρη ε, αυτή καθεαυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι αυτό εφικτό και επιθυμητό είναι η ερώτησή μου. Από εκεί και πέρα αναφερθήκατε στο ότι θα πρέπει να εξαρτόμαστε λιγότερο ε, ως προς την ασφάλεια των γραμμών προμήθευσής μας σε πόρους ενέργειας. Δηλαδή να εξαρτώμαστε λιγότερο από αγωγούς για παράδειγμα, γιατί εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό από αγωγούς για την, ε, τον ανεφοδιασμό μας σε ε, ενέργεια. Να εξαρτώμαστε λοιπόν λιγότερο από αγωγούς και περισσότερο από άλλες οδούς μεταφοράς και κυρίως θαλάσσιες οδούς αυτό θα διασφαλίσει ασφάλεια σε υψηλότερο βαθμό και αν ναι συμφιλιώνεται και συμβιβάζεται με τις επενδύσεις ε, και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το δίκτυο αγωγών ώστε να συνδεθεί με τις υπόλοιπες περιφέρειες και περιοχές του κόσμου όπως είναι η Μέση Ανατολή, η Ρωσία και η Βόρεια Αφρική. Άλλωστε, ε, προγραμματίζεται να δαπανηθούν πάρα πολλά χρήματα ε, στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη διασύνδεση της Ευρώπης και στο πλαίσιο της ενίσχυσης όλων αυτών των δικτύων. Και τέλος, ένα ερώτημα που απευθύνεται σε όλους σας. Τι επιπτώσεις θα έχει στη δική μας ασφάλεια το γεγονός ότι τώρα με την ε, οικονομική και δημοσιονομική κρίση στην ε, Ευρώπη αναδύονται άλλοι παίκτες, Κινέζοι και Ασιάτες, οι οποίοι αγοράζουν στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη. Π.χ. Ε, ένας προβλήτας στο Πειραιά έχει αγοραστεί από κινέζικη εταιρεία. Αγοράζουν λιμάνια λοιπόν σε ευρωπαϊκό έδαφος ε, εταιρείε από τη Σιγκαπούρη ελέγχουν άλλου είδου αντίστοιχε υποδομέ, λιμενικέ με πάρα πολλέ ε, και υψηλέ προοπτικές για την άνθεση του εμπορίου. Έχουμε όμως εκεί και περιορισμούς ως προς την αιρεσιμότητα, τους όρους με τους οποίους γίνονται όλα αυτά. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό το θέμα. Και τέλος, ε, ως προς τον αντινάβαρχο κύριο Φέλτ, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Χρειαζόμαστε πράγματι να δράσουμε μαζί και αν ναι, τι μας χρειάζεται για να το καταφέρουμε. Ποιες ικανότητες χρειαζόμαστε και θα πρέπει να επενδύσουμε για την οικοδόμηση αυτών των ικανοτήτων από πλευράς εξοπλισμού, επικοινωνιών αλλά και καλλιέργειας μιας άλλης νοοτροπίας, ενός νέου κλίματος. Ε, μου άρεσε πολύ η προσέγγισή σας για το ότι θα πρέπει να υπάρχει ευθύνη, αίσθημα ευθύνης για το μοίρασμα των ε, πληροφοριών, για την ε, διανομή τους. πού θα μπορούσαμε να επενδύσουμε με πιο ορθολογικό τρόπο για την ευρωπαϊκή διάσταση της θάλασσας κάτι το οποίο είναι πολύ πιο λογικό από το να αφήνουμε ε, το κάθε κράτος μέλος να μεριμνά από μόνο του, κάτι το οποίο δημιουργεί τον κίνδυνο επικαλύψεων. Και τέλος, αναφερθήκατε σε κάτι το οποίο είναι αλήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ε, επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Χρειαζόμαστε με την παγκοσμιοποίηση έναν πιο ρυθμισμένο κόσμο αν θέλετε και αυτό είναι κρίσιμης σημασίας, ζωτικής σημασίας. Έχει ε, παγκόσμια εμβέλεια. Με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι απειλές και με τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την ασφάλεια της θάλασσας έχετε την ε, αίσθηση ότι τελικά οι ΙΠΑ θα, συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική είναι η σύμβαση αυτή για το δίκαιο της θάλασσας. Ευχαριστώ. Ως ειδική εισηγήτρια έχετε ειδικά δικαιώματα και γι' αυτό ξεπεράσετε τα τρία λεπτά. Κύριε Χέλερ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και μας δίνει δυνατότητα να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτη. Επειδή υπάρχουν διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες, επιτρέπεται όλο και περισσότερα εμπορικά σκάφη να χρησιμοποιούν διάφορες ε, υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια αύξηση της ασφάλειας, αλλά τίθενται και λειτουργικά, νομικά θέματα. Πώς συνεργάζονται, για παράδειγμα, αυτές οι εταιρείες ασφαλείας με στρατιωτικές αρχές. διότι υπάρχουν διαφορετικά νομικά καθεστώτα και δυνατότητες παρέμβασης. Θα ήθελα να μας πείτε στην πράξη πώς έχει λειτουργήσει αυτή η ρύθμιση, έχει αυξηθεί η ασφάλεια στα πλοία, υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών των στρατιωτικών και αυτών των ιδιωτικών εταιρείων ασφαλείας. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τη χρήση αυτών των εταιριών. Και δεύτερον, Πολλές από αυτές τις εταιρείες δεν παρέχουν μόνο ασφάλεια, αλλά προσπαθούν αυτές οι εταιρείες να βοηθήσουν ούτω ώστε να μην αλλιεύουν σκάφη ε, από τα κράτη-μέλη, από τρίτα κράτη ε, σε περιοχές που δεν θα προεβλέπεται. Ε, έχει επιτευχθεί τίποτα στον τομέα αυτό. Τέτοιου τύπου θέλω να κάνω. Τώρα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρόκληση, η μέγιστη πρόκληση να απαντήσετε σε 6-7 λεπτά ο καθένας. Θα απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις Άρα θα επιλέξετε τις ερωτήσεις του δικού σας ενδιαφέροντος. Αν θέλετε μπορείτε να μιλήσετε και γερμανικά και πορτογαλικά ή να χρησιμοποιήσετε και άλλη γλώσσα πλην των αγγλικών. Ε, Θα είμαι σύντομος. Έχετε δίκιο όταν μιλάτε για τη μαύρη θάλασσα, όταν αναφέρεστε σε αυτήν. Η Τουρκία ε, είναι πλέον ιδιοκτήτης ε, τερματικών σταθμών πετρελαίου και καταβάλλεται προσπάθεια αποστολής πετρελαίου και στη Λιβύη, ακόμα από την περίοδο πότε έπρεπε να απομακρυνθεί ο Καντάφη. Ε, υπήρχε αυτός ο εμπορικός αποκλισμός δεν μπορώ να μιλήσω για τα ε, ρωσικά πολεμικά πλοία στη Συρία. Ε, αλλά υπήρξε μια κίνηση και προς το Λίβανο και θα ήταν σκόπιμο να δούμε τις εξελίξεις ως προς τις απειλές τις οποίες αναφέρθηκε η Άννα Γκόμες. Είναι πολύ δύσκολο ακόμα και να εικάσουμε αλλά σε σχέση με τις ε, πετρελαιοκυλίδες υπάρχει εγνωσμένος κίνδυνος και παρά την ε, ε, πολύ καλή εργασία που έχει γίνει στον τομέα αυτό με την άντληση πετρελαιοκυλίδων, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αντιμετωπιστεί το θέμα ούτε από την ακτοφυλακή, ούτε από τα πλοία στις υπεράκτιες περιοχές, διότι υπάρχουν πολλοί ε, φορείς που θέλουν να ε, περικόψουν το κόστος και αυτό είναι μία και από τις αιτίες δημιουργίας τέτοιων ατυχημάτων και γι' αυτό οι βιομηχανίες και οι φορολογούμενοι χάνουν δεκάδες εκατομμυρίων. Και αυτό βεβαίως τάσεται και κατά της ε, βιοπικιλότητας. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το επόμενα ε, το επόμενο ατύχημα, το μόνο που θα πούμε εκ των υστέρων είναι «Α, δεν το περιμέναμε». Αν υπήρχαν περισσότεροι τρομοκράτες και πιο έξυπνοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν και αυτό το τομέα διαφορετικά, ο οποίος είναι πολύ ευάλωτος. Αυτό που είναι ε, παράλογο είναι ότι υπάρχει μία εταιρεία από μία χώρα της ε, Βόρειας Ευρώπης η οποία μεταφέρει όπλα και πυρομαχικά σε πολύ ευαίσθητες περιοχές. Δεν ε, πρόσεξαν ιδιαίτερα τη διαχείριση αυτής της αποστολής και μέλη του προσωπικού κρατούνται από τους τρομοκράτες εδώ και πολλά χρόνια. Και ε, σε αυτή την περίπτωση και στο Μαυροβούνιο έγινε φόρτωση πυράβλων που έπρεπε να μεταφερθούν στο Βιετνάμ. Αυτή η εταιρεία είναι μια εταιρεία η οποία δυστυχώς είναι πολύ, ακολουθεί πολύ ε, επικίνδυνη πολιτική και πολλές φορές γίνεται μεταφορά ε, μιας, υπάρχει μια φόρτωση που μπορεί να αφορά πυράβλους ή και πυρηνικά. Και είδαμε πολλά τέτοια ατυχήματα μέσα σε αυτά τα κοντέινερ. Αυτοί οι κύριοι όμως μπορούν να ανοίγουν παραθυράκια και να κινούνται όπως θέλουν. Δυστυχώς ο θαλάσσιος τομέας δεν ελέγχεται επαρκώς σε σχέση με τις γήινες μεταφορές. Το Φεβρουάριο του 12 μετά τη σύραξη, μετά την απαρχή της σύραξης στη Συρία, ε, ο κατάλογος που είχε το ΝΑΤΟ των ε, επικίνδυνων μεταφορών, ή των ύποπτων μάλλον, που γνώριζαν και όλοι οι ομόλογοι, ενήχε ένα μόνο σκάφος, ένα πλοίο. και το πλοίο αυτό μεταφοράς όπλων προς την κυβέρνηση Ασάντ από ε, νιολογημένο στη Ρωσία πλοίο δεν ενεχόταν σε αυτό το κατάλογο. Γι' αυτό θέλω να πω, τι θέλω να πω με όλα αυτά. Είναι βάλωτος ο τομέας γιατί δεν ελέγχεται όσο οι εναέριες μεταφορές και οι ε, μεταφορές, ε, ε, δια τις, ε, οι οδικές μεταφορές. Ο κύριος Πίτα ελέχθη, τι μπορούμε να κάνουμε έμπρακτα ως συνέχεια. Μεγάλη πρόοδος μπορεί να επιτελεστεί μετά την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλεια του 2003 που αναφέρθηκε και στη θαλάσσια ασφάλεια. Από το 2003 μέχρι σήμερα έχει εξελιχθεί η κατάσταση, αλλά πολύ ταχύτερα από ότι η αρχική μας σκέψη ως προς τη θαλάσσια ασφάλεια. Αν δούμε τον κόλπο της Γουινέας, έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση που δεν είχε καμία σχέση με το 3. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει πειρατεία που αφορά και την Νότια Αμερική και την Αφρική και η πολιτική η εξέλιξη στο Σαχέλ δείχνει ότι η τρομοκρατία επίκειται και σε αυτή την περιοχή. Υπάρχουν μεγάλοι κλειδονισμοί και μία πτητικότητα στην εξέλιξη και στα σύνορα σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, με τα καύσιμα γενικότερα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να κινηθούμε τάχιστα. Θα απαντήσω στα πορτογαλικά για την ακτοφυλακή, την ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Χρειάζεται η ευρωπαϊκή αυτή ακτοφυλακή, πρέπει να δημιουργηθεί είναι ένα θέμα πολύ σχηδές όμως, διότι τα πολιτισμικά πλαίσια είναι διαφορετικά σε σχέση με την εθνική εποπτεία, θέματα εθνικής εποπτείας στα παράκτια. Υπάρχει η αρχή του πολεμικού ναυτικού που εποπτεύει τα παράκτια, ιδιαίτερα στη Γαλλία, και αυτό ισχύει και στην Πορτογαλία. Υπάρχει ένα διαφορετικό πρότυπο ακτοφυλακή σε άλλες χώρες, όπως στην Ολλανδία. Υπάρχει επίσης ένα άλλο πρότυπο που αποτελεί σύμιξη των δύο, δηλαδή πολεμικού και ε, πολιτικού ναυτικού. Και Υπάρχει σωρία οργανισμών εποπτείας των παρακτήων που δεν μπορούν να συντονιστούν μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι το σημείο κίνησης είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Εάν σκεφτούμε όπως τα κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι κατά την σύνταξη της πράσινης ε, βίβλου για την ε, ολοκληρωμένη ναυσιπλοεία των κρατών μελών, όλα τα κράτη-μέλη, εκτός πλην ενός, μιλώ για τα παράκτια κράτη, δεν ήθελαν να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Πλην ενός κράτους. Μία ενιαία ευρωπαϊκή ακτοφυλακή μεταξύ αυτής της ενιαίας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής και του τωρινού προτύπου υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ε, μία δομή τύπου ΝΑΤΟ. Γιατί εκεί υπάρχει μία ενιαία δομή με ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ διαφόρων χωρών. Γι' αυτό υπάρχουν περιθώρια για εξέλιξη. Δεν μπορούμε όμως να μην διαθέτουμε ικανότητες διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ εθνικών ακτοφυλακών. Και ως προς το τελευταίο ε, ερώτημα σε σχέση με τις οδούς ενέργειας και λιγότερους αγωγούς Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 90, η θαλάσσια μεταφορά ορυκτών καυσίμων αποτελούσε ένα θέμα ταμπού. Μετά τα ατυχήματα και τις πετρελαιοκυλίδες ε, στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 80 και 90 υπήρξε μεγάλη δημόσια κατακραυγή για τις θαλάσσιες μεταφορές. Τότε αποφασίστηκε ότι ότι μόνο τα δίκητα τάνκερ θα μπορούσαν να διαπλέουν την Ευρώπη. Και υπήρχε μια προθεσμία, μια καταληκτική ημερομηνία του 2009. Και τότε όλα τα τάνκερ ε, που μετέφεραν πετρέλαιο ήταν δίκητα. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Όταν ο Επίτροπος Πίμπαλξ ήταν υπεύθυνος για θέματα ενέργειας, έλεγε στα κράτη-μέλη ότι χρειαζόμαστε περισσότερα τερματικά LNG. Είχαμε περίπου 20, κάτι το οποίο είναι παράλογο γεωπολιτικά διότι η εξάρτησή μας από τους αγωγούς είναι πολύ μεγάλη. Όσο περισσότερο ε, κανείς βρει εναλλακτικές οδούς, τόσο καλύτερη προμήθεια έχει. Επίσης, σε σχέση με το φυσικό αέριο, βλέπουμε ότι κινούμεθα σε αγορές spot όπου οι, οι τιμές συνάδουν ή πλησιάζουν τις τιμές του πετρελαίου. Γι' αυτό η ενεργειακή προμήθεια έχει μεγάλη σημασία και σε επίπεδο ασφάλειας, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει να ξαναδούμε την ενεργειακή μας πολιτική, την ενεργειακή προμήθεια στην Ευρώπη για να αποφύγουμε τα πρόσφατα ατυχή γεγονότα που γνωρίσαμε στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη όπου δεν υπήρχε ε, δυστυχώς θέρμανση. Ευχαριστώ. Τώρα ο αντινάβαρχος ο κύριος Φέλντερ. Με συγχωρείτε, ε, θα επιχειρήσω τώρα να μιλήσω πιο αργά, τουλάχιστον στην αρχή. Θα επιχειρήσω να απαντήσω ορισμένες ερωτήσεις ε, για τις οποίες νομίζω ότι κάτι μπορώ να πω. Καταρχάς, να τονίσω πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Και από εκεί θα δούμε τι χρειαζόμαστε ως περισσότερες δυνατότητες. Νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά ναυτικά έχουν πολλές δυνατότητες για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τις απειλές επί των οποίων όλοι συμφωνούμε. Έχουμε δυνατότητα. Αυτό που μας λείπει και κατέστη ήδη σαφές είναι ότι δεν υπάρχει η, η βούληση να χρησιμοποιήσουμε από κοινού και να μοιραστούμε τις δυνατότητες. Pooling and sharing. Πρέπει να γίνει σωστά. Και αν γίνει σωστά, αυτό σημαίνει ότι οι χώρες που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να εκχωρήσουν ένα τμήμα της κυριαρχίας τους στην Ένωση. Αυτό πρέπει να αποφασίσει. Εσείς θα αποφασίσετε ποια αρχή, ποια αρχή θα αναλάβει αυτό το τμήμα της κυριαρχίας. Αλλά η πλήρης και σωστή απάντηση είναι ότι αυτό το pooling και sharing θα είναι βοηθητικό βέβαια, αλλά ε, δεν αρκεί εάν οι πολιτικοί το θεωρούν μόνο ως μέσο εξοικονομήσεων. Ένας δεύτερος τομέας που θεωρώ ότι είναι ζωτικός για πιο έντονη συνεργασία και για τους τρεις τομείς, τομείς ενεργική, ασφάλεια και άμυνα και επανέλθω σε αυτό που είπατε, είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Αν σκεφτούμε ότι και εντός των κρατών μελών αλλά και στην Κομισιόν υπάρχει πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, την αμοιβαία πληροφόρηση και πολλές φορές φτιάχνουμε φράγματα αντί να φτιάχνουμε δυνατότητες επικοινωνίας και στον πολιτικό και στον στρατιωτικό. Εδώ υπάρχει έλλειψη κυρίως στον πολιτικό όμως τομέα, γιατί οι στρατιώτες έχουν συνηθίσει να συνεργάζονται. Η Κομισιόν πρέπει να δημιουργήσει μια κοινή δυνατότητα ανταλλαγής προφοριών. Αυτή είναι μια πολύ ρεαλιστική πρόταση και πρέπει να τύχει περισσότερης πολιτικής υποστήριξης. Και πρέπει να καταστεί σαφέ, γιατί τώρα δεν είναι σαφές, ότι αυτή η συνεργασία θα βοηθήσει. Ποιε είναι τώρα οι ρωσικές προθέσεις. Η Ρωσική Ομοσπονδία αποφάσισε ότι θα έχει μόνιμη ναυτική, πολεμικού ναυτικού δηλαδή παρουσία, στην ε, Μεσόγειο. Αυτό ο στόλο υπάρχει. Δεν ξέρουμε τώρα ποια λιμάνια θα χρησιμοποιήσει, αλλά υπάρχει. Η πληροφόρησή μου είναι ότι προτίθενται να έχουν μόνιμα πολεμικό ναυτικό και στον Ατλαντικό και στον Ινδικό. Είναι σαφής λοιπόν η κατεύθυνση και νομίζω ότι απήντησα. Λοιπόν, βεβαίως αυτό έχει να κάνει με τη δική μας πολιτική γειτονία. Αλλά είναι σαφές ότι θα γίνει αυτό. Υπενθυμίζω, η Ρωσική Ομοσπονδία ήδη έχει συμμετάσχει και σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ για ένα διάστημα. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχει και τέτοια συνεργασία στη Μεσόγειο για συγκεκριμένε δραστηριότητε. Γιατί να μην καλέσουμε τη Ρωσική Ομοσπονδία για να κάνουμε από κοινού ασκήσει. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε εντάσει, διότι υπάρχει περισσότερη αλληλοκατανόηση και συμφωνούμε σε κοινού στόχου. Και γιατί, για παράδειγμα, να μην αξιοποιήσουμε το καλό παράδειγμα της επιχειρήσης Αταλάντα. Δηλαδή, να μην ε, οδηγήσει αυτή η εμπειρία ε, να αναλάβουμε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και την ηγεσία του Unifil. Έχουμε τα μέσα να το κάνουμε. Υπάρχουν κράτη-μέλη που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια πλατφόρμα. Υπάρχουν πολλά λοιπόν που ήδη σήμερα μπορούμε να κάνουμε, όπου έχει τις δυνατότητες η Ένωση. Για την εφαρμογή αυτών των δυνατοτήτων όμως, πολλά κράτη τονίζουν ότι δεν τους επιτρέπουν ε, τα οικονομικά τους να ε, συμβάλλουν μέσω σκαφών και αεροσκαφών σε αυτές τις προσπάθειες. Αυτό πρέπει να επιληθεί με διμερείς και πολυμερείς επαφές. Για την θάλασσα της Νότιας Κίνας. Υπάρχει μεγάλη ένταση εκεί και οι αναλυτές από την περιοχή υπολογίζουν ότι η πιθανότητα πολέμου θαλάσσιων συγκρούσεων είναι 60%. Την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχα σε μια συζήτηση όπου ήταν πολύ σαφής οι Κινέζοι, ήταν πολύ σκληροί στις ε, δηλώσεις, του, στις δηλώσεις τους κατά της Ιαπωνίας. Υπάρχει μια σύγκρουση. Και τέθηκε το ερώτημα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τέτοια εμπειρία για λύση τέτοιων συγκρούσεων και για μείωση των εντάσεων, για αποκλιμακώσεις, γιατί να μην προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ουδέτερο διαμεσολαβητής να βοηθήσει τα κράτη αυτά, τα οποία είναι κράτη με τα οποία έχουμε ε, πολλά κοινά στοιχεία, πολύ στενέ σχέσει. Γιατί και με την Κίνα έχουμε πολύ στενέ σχέσει. Γιατί λοιπόν να μην επιδιώξουμε να βοηθήσουμε να υπάρξει αποκλιμάκωση. Εάν υπάρξει φυσικά η πολιτική βούληση της Ένωσης να εμπλακεί, να κάνει μια προσφορά προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα τώρα για τις υπηρεσίες ασφαλείας στα σκάφη, τις υπηρεσίες ιδιωτικής ασφαλείας. Βεβαίως, από τότε που υπάρχουν ε, ιδιωτικοί ε, άνδρες ασφαλείας στον Ειδικό Ωκεανό, δεν έχουν μειωθεί οι επιθέσεις, αλλά έχουν μειωθεί οι επιτυχεί επιθέσεις και μάλιστα ουσιοδό. Αυτό είναι το καλό νέο. Αλλά πρέπει να πω, και είναι προσωπική μου άποψη, ότι η λύση αυτή δεν είναι σίγουρα η καλύτερη. Δεν είναι δυνατόν να εχωρούμε τις αρμοδιότητες ασφαλείας και χρήσεως όπλων κυρίως χρήσεως όπλων. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Και ξέρω ότι πολλοί Γερμανοί και άλλοι Ευρωπαίοι εφοπλιστές θεωρούν σαφώς ότι θα ήταν καλύτερα να είναι αστυνομικοί ή στρατιώτες στα πλοία μας. Ένα είναι σαφές. Εάν ε, σκοτώσει κάποιον ένας ε, άνδρας ιδιωτικής ασφαλείας, ένας ιδιωτικός φρουρός, τότε την ευθύνη την έχει ο πλοίαρχος, όχι ο ιδιωτικός φρουρός. Δεν είναι λοιπόν η καλύτερη λύση αυτή. Και κάτι ακόμη, τελευταίο, για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, για την Σύμβαση των ΗΠΑ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ούγκλος. Αυτό το Δίκαιο της Θάλασσας προέκυψε μέσω μιας διαδικασίας που δεν ε, ε, λαμβάνει υπόψη τις ε, ασύμετρες απειλές που υπάρχουν σήμερα. Άρα αυτές τις ασύμετρες τρομοκρατικές και άλλες εγκληματικές ενέργειες και απειλές δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει γιατί δεν τις προέβλεπε. Σημαντικό λοιπόν είναι να ανεπτυχθεί περαιτέρω το δίκαιο αυτό και πρέπει να συμμετάσχει εντόνως η Ένωση και λοιπόν μια στρατηγία της θάλασσας για την αυσιπλοεία θα ήταν μια καλή αρχή για να μπορέσουμε να εργαστούμε ορθώς και εντόνως στον τομέα αυτό και το δεύτερον, αμφιβάλλω ιδιαίτερα, εάν η Ινδία, η Βραζιλία και η Κίνα θα θελήσουν να μην συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Διότι, βεβαίω, θα πούν ότι θέλουν να συμμετάσχουν στο μέλλον πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν και δεν είναι μειονέκτημα αυτό. Αντίθετα, αυτό θα ήταν ε, θαυμάσιο προτέρημα αυτή τη διαδικασία να συμμετάσχουν και αυτέ τι χώρε αυτή εξ αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους. Φυσικά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για τη θαλάσσια διάσταση της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας όταν θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε την έκθεση της κυρίας Γκόμες. Ευχαριστώ όλους. Ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας.